συνέβησαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ευρωβουλευτά για αυτή την παρέμβασή σας. Φυσικά σε τέτοιου είδους σημαντικά γεγονότα αν έχουν συμβεί με αυτόν τον τρόπο σίγουρα θα τύχουν τις προσοχή μας θα ασχοληθούμε με αυτά σας ευχαριστούμε για την παρατήρησή σας περνάμε τώρα στις ε, τακτικές εργασίες μας σύμφωνα με τις ε, κοινοβουλευτικέ ομάδες προτείνουμε οι συζητήσεις ε, για απόψε να έχουν ως εξής Δευτέρα απόψε Πρώτον, θα έχουμε τις προφορικές ερωτήσεις ε, για την ευρωπαϊκή πολιτική αλίας, για τον τομέα της αλίας και την κρίση στον τομέα αυτό, σαν αποτέλεσμα της άφησης των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων του πετρελαίου. Και δεύτερον, η έκθεση του κυρίου Χεκμακ ε, για το φάσμα, ε, το ραδιοφάσμα όσον αφορά την πολιτική μας για τεχνικούς λόγους έχει σχέση και με την παρουσίαση και συμμετοχή επιτρόπων. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Αυτή η αλλαγή αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν έχουμε τίποτα για την Τρίτη, δεν υπάρχουν αλλαγές. Για την Τετάρτη στη συνέχεια. Για την Τετάρτη υπάρχει κάτι που αφορά τον κύριο Σπερώνη. Ο κύριος Σπερώνη θα, θα εξηγήσει όσον αφορά την συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Ζητήθηκε από πλευρά της, ε, για την Επίτροπο για την, ε, και είπα το εκπρόσωπο να συμπεριληφθεί η κατάσταση στην ε, Συρία και η κατάσταση της κοπτικής κοινότητας χριστιανών στην Αίγυπτο. Είναι ένα αίτημα το οποίο αφορά την Τετάρτη, την πρωινή συζήτηση την Τετάρτη στις 9 η ώρα με την Λέδη Άστον, είπα το εκπρόσωπο. Ο συμπρόεδρος Περών έχει τον λόγο για να εξηγήσει το αίτημα παρακολουθεί. Κύριε Πρόεδρε, δεν θελήσαμε να προτείνουμε τροποποιήσεις επί της ουσίας στην ημερήσια διάταξη. Δεν θέλαμε ούτε να την επιβαρύνουμε ούτε να αντικαταστήσουμε. Διευρύνουμε όμως, η πρότασή μας είναι να διευρύνουμε το θέμα στο οποίο μόλις εσείς αναφερθήκατε και ζητάμε ουσιαστικά να προσθεθεί στο υποσυζήτηση θέμα για το θέμα του Αστραφ και το θέμα ευρύτερα της χριστιανικής μειονότητας, της κοπτικής χριστιανικής μειονότητας κυρίως στην Αίγυπτο. Πρόκειται για μια μεγάλη ευαίσθητη ζώνη και ένα θέμα το οποίο έτσι και αλλιώς καλύπτει ότι έχει σχέση με τις μειονότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα ήθελε να εκφραστεί θετικά υπέρ αυτού του θέματος, ο κύριος Γκόλνης. Θετικά παρακαλώ, είστε υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά και είμαι υπέρ αυτού του αιτήματο. Σας είχα ζητήσει το λόγο και για την ημερήσια διάταξη της ημέρας Τρίτης. Θα μου, δώσετε, θα μου δώσετε τώρα τη δυνατότητα να μιλήσω ή μετά το τέλος της παρέμβασης περώνει. Κοιτάξτε, πρώτα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για την Τετάρτη που έχουμε αρχίσει να συζητάμε. Ο κύριος Μπεντίτ θα, θα μιλήσει υπέρ, όχι, είναι κατά της συμπερίληψης αυτής. Ο κύριος Μάουρο είναι υπέρ. Ο κύριος Μάουρο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με το αίτημα του κυρίου Σπερώνη Θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συγκρούσεις που εμπλέκουν και την κοπτική κοινότητα είναι ένα μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο δείχνει τους κινδύνους αυτού του οποίου συμβαίνει στην Αίγυπτο. Το αίτημα πρέπει να υποστηριχθεί λοιπόν. Το θέμα δεν είναι εμείς να υπερασπίσουμε κάποιες διαδηλώσεις υπέρ της ταυτότητας μιας συγκεκριμένης θρησκευτική μειονότητας. Νομίζω ότι εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω της δήλωσης την οποία θα πρέπει να κάνει η κυρία Άστον πρέπει να δείξουμε το ενδιαφέρον μας. Κύριο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι εξεπλάγετε από αυτά τα οποία συνέβησαν στην Αίγυπτο. Πρέπει να είμαστε όμως λογικοί. Έχουμε έξι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με την κυρία Άστον. Το θέμα της Συρίας, το θέμα του Ασράφ, έχουμε την έκθεση Γουαλτιέρη, έχουμε την έκθεση Αλμπερτίνη, έχουμε την έκθεση ε, της Ευρώπης ε, ε, σφαιρικού παίκτη στα Ηνωμένα Έθνη Όλα αυτά λοιπόν είναι πολλά. Πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσει αυτή την κατάσταση στην Αίγυπτο, περιλαμβάνοντας όλα όσα έχουν συμβεί ανάμεσα στις θρησκευτικέ μειονότητες, κοινότητες μάλλον. Να υπάρξει μια έκθεση πρωτοβουλίας και μια συζήτηση με την κυρία Άστον σε έφθετο χρόνο, αλλά η συζήτηση να είναι πραγματική. Άμα πραγματικά προσθέσουμε ένα έκτο σημείο, τότε μόνο ένας θα μιλήσει για το θέμα, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, έξι θέματα στη συζήτηση με την Βαρόνι Άστον δεν θα συγκεντρώσετε την προσοχή ε, του κοινού και των συναδέλφων. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να επιβαρύνουμε ε, την συζήτηση της Τετάρτης το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κον Τώρα θα συνεχίσουμε με, τις, με την ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ της προτάσεως την οποία μόλις έκανε ο κύριος Περόνη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι κατά. Κοιτάξτε, ε, θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πάρτε τις κάρτες σας, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Περιμένω, ψηφίσατε όλοι. Καλώς. Τέλος της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ε, γίνεται δεκτή η πρόταση την οποία έκανε ο κ. Σπερώνη και θα προσθεθεί το θέμα αυτό στην συζήτηση ε, την Τετάρτη το πρωί. Κύριος Γκόλνης έχει δει το λόγο εκ νέου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε πάλι το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Η διάσκεψη των Προέδρων προβλέπει για αύριο, για αύριο Τρίτη, μια ψηφοφορία για την πιθανή άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας. Δεν θα μπω στην ουσία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Θα ήθελα όμως, σχετικά με την ημερήσια διάταξη καθεαυτή, να πω ότι με αρνητικά και με πολύ αρνητικά γιατί ότι δεν προβλέπεται συζήτηση και δεν θα μου δοθεί δυνατότητα ούτε μέσα σε ένα-δυο λεπτά να παρουσιάσω τη θέση μου. Νομίζω ότι η θέση μου θα είχε κάποιο ενδιαφέρον. Ο εισηγητής επανέρχεται στην προηγούμενη υπόθεση, την υπόθεση που είχε προκαλέσει η κυρία Βόλης, που είχε οδηγήσει στην άρση της κοινοβουλευτικής μου ασυλίας, κάτι το οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε καταδικάσει σαν θέση. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν είναι διαστεκαστικό δεν πρόκειται για κάτι το διαδικαστικό. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Γκόλνης. Επανέρχεται ο ήχος του κύριου Γκόλνης. Λοιπόν, εγώ ζητάω ε, δύο λεπτά. Θέτω ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θέλω δύο λεπτά για να υπερασπίσω την τιμή μου. Ακούστε με, έχω δικαίωμα σε κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν να σεβαστείτε έστω και για μία μέρα τα δικαιώματα, εν περιπτώσει, της υπεράσπισης ή πρέπει να πάμε στη Γουατεμάλα και την Ινδονησία για να προασπίσουμε τα πολιτικά μας δικαιώματα. My postępujemy, panie panie kolego my postępujemy zgodnie z zasadą... Αγαπητέ συνάδελφε Γκόνης, εμείς θα προχωρήσουμε και θα πράξουμε ανάλογα με αυτά τα οποία προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 8. Άρθρο 7, παράγραφος 8. Το άρθρο αυτό συγκεκριμένα είναι ξεκάθαρο. Λέγει ότι το θέμα το οποίο θέσατε έπρεπε να το είχατε θέσει μία ώρα πριν από την αρχή της συγκεκριμένης αυτής συνεδρίασης. Αναφέρομαι στο άρθρο 7 παράγραφος 8. Συνεπώς λοιπόν επανερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με την Τετάρτη, λέει ο κ. Κονπεντίτ. Και να πω κάτι για την ημερήσια διάταξη της ημέρας Τετάρτης. Κοιτάξτε, η διάσκεψη των Προέδρων, λέει ο κ. Κονπεντίτ, προβλέπει για την Τετάρτη το απόγευμα μια συζήτηση για τις προτάσεις της Ιταλικής και της Γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με την προσωρινή διακοπή της σύμβασης Σέγγεν. Την τρίτη το απόγευμα διορθώνει ο κ. Κονμπεντήτ Λοιπόν, είχε αποφασιστεί επίσης ότι ο κύριος Μπαρόζο θα πρέπει να είναι παρόν στη συζήτηση αυτή. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του Πρόεδρου της Επιτροπής. Γιατί, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πήρε θέση μετά από τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις δύο μεγάλες προσωπικότητες, τον κύριο Μπερλουσκόνη και τον κύριο Σαρκοζή, ήταν ο Πρόεδρος ο κύριος Μπαρόσο. Ενώ οι επίτροποι του εξέφασαν διαφορετικές θέσεις. Θυμίζω ότι στην Επιτροπή, ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τη θέση την επίσημη της Επιτροπής. Γι' αυτό εμένουμε στην παρουσία του κυρίου Μπαρόσο την τρίτη του απόγευμα στις 3 το μεσημέρι. Συγγνώμη για την πέρδεψα την τρίτη και την τετάρτη. Θα το ελέγξω λέει ο πρόεδρος. Κύριε Συμπρόεδρε θα το ελέγξω. Θα το ελέγξω αμέσως. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα το κοιτάξω. Υποθέτω ότι θα είναι παρόν ο κύριος Μπαρός. Υποθέτω λέω, αλλά άλλη πληροφορία δεν έχω. Θα το ελέγξω όμως. Θα κάνω μια ειδική κίνηση χάρης ε, για χάρη σας. Uh, colleague Gianni, if I could ask Mr. Vice President. Great. The next point is... Λοιπόν, το επόμενο σημείο... We must change ourselves. Ε, είναι γραμμένο στα Ιταλικά, οπότε προφανώς πρέπει να μεσολαβήσει μια κάποια αλλαγή. Ehm, λοιπόν, γεια σας. Ε, θεωρούμε δεδομένη την υιοθέτηση της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Συζήτηση για την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κρίση